przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego jest... Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Το πρώτο θέμα είναι της ημερήσιας διάταξης. Είναι η έκθεση της κυρίας Καρνιέτε, διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά καθώς επίσης η έκθεση του κυρίου Ντεκάμπος εν η αγορά των Ευρωπαίων πολιτών εν η αγορά για τις επιχειρήσεις που έχει κοινή συζήτηση βεβαίως Σίλβιο Μπουσόη και δημόσια σύμβαση δήλωση της Επιτροπής εγώ απευθύνω το καλώς ορίσατε στον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ καθώς επίσης και την εκπρόσωπο της Προεδρίας, την ε, Υπουργό κυρία Γέρη. Πρώτα θα δώσω το λόγο στους τρεις εισηγητές και πρώτα η κυρία Σάντρα Καρνιέτη. Madame Kalniete. Ah, Mr. President, sorry. I... Με συγχωρείτε Πρόεδρε. Μέχρι να ακούσω τη μετάφραση της ε, εκφώνησής σας, καθυστέρησα. Πιστεύω, Πρόεδρε, ότι αν θέλουμε να πιστεύουμε στην ιστορική αγορά, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραματίσει έναν ηγετικό ρόλο. Αυτό είναι το κύριο, το κύριο καθήκον μας. Έτσι λοιπόν με την ε, υποστήριξη τόσο του Συμβουλίου όσο και ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να βοηθήσουμε στην ε, καλύτερη ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Υπάρχει ανάγκη να προβάλλουμε νέες ιδέες για την ανάπτυξη, την οικονομική, τη δημιουργία νέων θέσεων την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς μας αλλά όσες ιδέες και αν προβάλλονται μερικές φορές παραμένουν μόνο στα λόγια. Γι' αυτό θα πρέπει πλέον να αναλάβουμε δράση. Γι' αυτό ζητούμε με το ψήφισμα από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνε τους και να προχωρήσουν και σε νομοθετικό επίπεδο και σε χάραξη πολιτικής για την προαγωγή της εσωτερικής αγοράς. Με τις εκθέσεις μας δίνουμε σαφείς ενδείξεις και ορίζουμε σαφή ορόσημα για το τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις συγκεκριμένε δράσεις. Μια κοινή ψηφιακή αγορά και, δικαίωμα, και προστασία των δικαιωμάτων του παραγωγού, η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, παροχή υπηρεσιών, κίνηση κεφαλαίων, φορολογία στην εσωτερική αγορά ενιαία και πρέπει τα κράτη-μέλη να επιτελέσουν το καθήκον τους με βάση τα όσα ορίζει ήδη η νομοθεσία ε, και υπό την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, θα πρέπει για να αποτραπεί ο κατακαιρματισμός της ιστορικής αγοράς να πάυσει ο προστατευτισμός που ακόμη υφίσταται. Τρίτον, θα πρέπει να μειωθούν ε, ε, τα τέλη των ε, συναλλαγών στα χρηματοπιστικά και εδώ ζητούμε συγκεκριμένη τιμολόγηση ε, διακύμανση των τελών με βάση συγκεκριμένα και σαφή κριτήρια στις ε, ηλεκτρονικές συναλλαγές και επίσης δυνάμει της συνθήκης Λισαβόνας θα πρέπει να συμμετέχουν ε, στην προετοιμασία των ε, νέων εξελίξεων και μέτρων και οι ομάδες των φορέων που αφορά αυτή η νομοθεσία και των διαφόρων παραγόντων. Πιστεύω ότι θα πρέπει το ψήφισμα να υιοθετηθεί, Προέδρε, έτσι ώστε να προχωρήσουμε, να βοηθήσουμε στην προαγωγή της εσωτερικής αγοράς. Η δουλειά αυτή δεν έχει φτάσει στο τέρμα τη. θα συνεχιστεί ασφαλώς για να καταστεί κινητήριος μοχλός της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και της ε, ανάπτυξη τη η εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, θαυμάσια οργανωμένη ομιλία σας. Ακολουθεί ο κύριος Αντώνιο Φερνάντο Κορέα Κάμπος. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε στο αίτημα τη Επιτροπή για να υπάρξουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόθεση της νέας αγοράς μέσω της παρούσας έκθεσης και των εκθέσεων που γενικότερα συζητούμε σήμερα. 19 προτάσεις προτάθηκαν από τις ομάδες σε ό,τι αφορά τα κριτήρια της ενιαίας αγοράς χρησιμοποιώντας μια σειρά ε, προτεραιοτήτων καταρχά την αύξηση της κινητικότητας των πολιτών με αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των, του, του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής ταυτότητας ε, ε, προσόντων και μέτρηση της κινητικότητας, της στην Ένωση. Δεύτερη, ε, ο, έλεγχος των, ο έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της αγοράς. Εφαρμογή τρίτων του κανονισμού του roaming μέχρι τον Ιούνιο του 2015, περιορίζοντας τις τιμέ του roaming, ούτω ώστε το κοινό και οι επιχειρήσει να πληρώνουν λιγότερο. Τέταρτον, πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές, τραπεζικές υπηρεσίες με μεγαλύτερη διαφάνεια. Και πέμπτον, ε, κατάργηση των εμποδίων των των εργαζομένων για να μπορέσουν να έχουν πλήρω τα δικαιώματα συνταξιοδότηση. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά. Ε, ήταν πολύ πιο δύσκολο ωστόσο, πολύ πιο δύσκολο ωστόσο να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην, να χτυπήσουμε την κόποση της ενίας αγοράς όπως αναφέρθηκε στην έκθεση Μόντι και να υπάρξει μια περιεκτική προσέγγιση για, την, για να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες του πληθυσμού που, ε, πρέπει να, που εντοπίζονται στην έκθεση Γκρέκ και που εγκρίθηκε πέρσι το Μάιο. Αναγνωρίζουμε την, ε, αναγνωρίζουμε βέβαια τις προσπάθειες της Επιτροπής ΙΜΚΟ για να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση και στις τρεις εκθέσεις του Κοινοβουλίου και οι τρει συνιστώσει, επιχειρήσει, πολίτε και διακυβέρνηση, θα πρέπει να προχωρήσουν ταυτόχρονα για να πετύχουμε μια ανταγωνιστική εσωτερική αγορά με έξυπνη ανάπτυξη και που θα είναι βιώσιμη και θα επιτρέψει στου Ευρωπαίου να είναι στο κέντρο τη ανησυχία τη αγορά αυτή. Αναγνωρίζουμε επίση ότι ο πολλαπλασιασμό πρωτοβουλειών τη Επιτροπή στο ζήτημα αυτό, η Ευρώπη 2020, η πολιτική για τη βιομηχανία και η Ευρώπη τη καινοτομία, μπορεί να οδηγήσουν στο να χάσουμε την εστίαση και την μείωση της ιδέας μας για την ανάγκη ε, ανανέωσης της εσωτερικής αγοράς που πρέπει να είναι προσπελάσιμη και κατανοητή στους πολίτες. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Ήταν δύσκολο να πετύχουμε συμφωνία σε δύο ζητήματα κυρίες και κύριοι. Πρώτον, σεβασμός των κοινωνικών αξιών και δικαιωμάτων. Χρειάστηκε να υπάρξει ε, η δεξιά και οι φιλελεύθεροι δεν ήθελαν να, δεχθούν μια πλήρη διαφύλαξη των κοινωνικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων για να μην πνιγούν οι Ευρωπαίοι στην απλή λογική της αγοράς στο μέλλον. Επίσης, λυπούμαστε γιατί δεν έγινε δεκτή ως προτεραιότητα η αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Δεύτερον, η διαφύλαξη των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ε, που, το, που έπρεπε να βγει από τη λογική της αγοράς με μείωση των δημοσι... με μετατροπή των δημοσίων υπηρεσιών όχι σε μονοπόλια ή ολιγοπόλια ε, ειδικά σε τομείς όπως η παροχή ύδατος, οι μαστικές μεταφορές κλπ. Δεν πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να θεωρηθούν ως απλές υπηρεσίες αγοράς και ταυτόχρονα προσπαθώντας να διαφυλάξουμε τις κοινωνικές αξίες και τις αρχές της αλληλεγγύης που θα πρέπει να υπερισχύσουν στην απλή λογική της αγοράς. Υπήρξαν αμφιβολίες και αντι Ρίσεις από πλευράς διαφόρων ομάδων της δεξιάς του Κοινοβούλιο που δεν δέχονται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά και λένε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις του άρθρου 14 και του πρωτοκόλλου 26 της συνθήκης. Η ομάδα μου απέσχε στην τελική ψηφοφορία για τις, τρες, για τις τρεις εκθέσεις στην Επιτροπή, διότι δεν υπήρξε καμία πραγματική πρόοδος στην κοινωτική διάσταση της εσωτερικής αγοράς παρότι το κείμενο είχε πολλές θετικές προτάσεις που βελτίωσαν, που βελτίωσαν. Οι τελικές τροπολογίες ωστόσο που, που, που, που, προτάθηκαν ε, από τις επιτροπές βελτίωσαν το αντικείμενο. Τελικό αποτέλεσμα είχαμε 266 τροπολογίες, ε, γνωμοδοτήσεις από πέντε διαφορετικές επιτρεπές. Οι συζητήσεις ήταν χρήσιμες. Ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές, Χόχενστάιν, Κρόιτσμαν, Χάρμπορ, Τούρνεν και Τριανταφυλλίδη, καθώς και τους συντονιστές των ομάδων για την παραγωγική πολιτική και το πνεύμα συνεργασίας που επέτρεψαν να ολοκληρωθούν οι οι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ ιδίω τον κύριο Χάρμπορ για το όραμα που έδωσε στι εργασίε τη Επιτροπή και τη διάρκεια του τετραμήνου που δουλεύαμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Έξι λεπτά είχατε στη διάθεσή σα. Σα έμεινε ένα λεπτό λοιπόν που θα χρησιμοποιηθείτε αργότερα στις τελικές παρατηρήσεις. Το ίδιο ισχύει για τον κύριο Κρίστιαν Σίλβιου Μπουσόη. Έξι λεπτά τέσσερα λεπτά στην αρχή και δύο λεπτά για τελικές παρατηρήσεις. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, η ιστορική αγορά είναι ασφαλώ μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει και μια από τι κυρίε δυνάμει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε όλοι να είμαστε υπερήφανοι. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πούμε ότι η ιστορική αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η ιστορική αγορά απέδειξε σε το χρόνο τα πλεονεκτήματά τη και για τον καταναλωτή αλλά και για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και έχει συμβάλει στην οικονομική μας ανάπτυξη. Πλην όμω, διαπιστώνεται μία κόπωση και στην ολοκλήρωση και στη λειτουργία τη ιστορική αγορά το τελευταίο καιρό και γι' αυτό χρειαζόμαστε νέα όθηση για την ιστορική αγορά. Χρειάζεται δηλαδή να τις ξαναδώσουμε ε, να ξαναβρεθεί η εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά για τον Ευρωπαίο πολίτη. Χρειαζόμαστε μια νέα αρχή. Εκτιμώ ιδιαίτερω τι ε, προσπάθειε Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου και ιδιαίτερω του κυρίου Μπαρνιέ, του κυρίου Επιτρόπου, τον οποίο για άλλη μια φορά συγχαίρω για τη στράτευσή του, για την επιμονή του και τι προσπαθίε του για την ε, παραπροώθηση τη εσωτερική αγορά Μα έχει προτείνει λοιπόν ένα φιλόδοξο αλλά και ταυτόχρονα απαραίτητο όσο και ρεαλιστικό πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ξαναδώσει πιστεύω την όθηση στην ε, εσωτερική αγορά. Είμαι πεπισμένο ότι αν ε, τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά θα καταστήσουν την εσωτερική αγορά πιο ελκυστική για του ε, καταναλωτέ και για τα εμπορεύματα. Και έτσι θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση μια εσωτερική αγορά. Αγαπητοί συνάδελφοι στα αγγλικά, είναι καθήκον αυτό το οποίο είχα να επιτελέσω καθόλου ε, ευτελές ή εύκολο. Ε, έχουμε δηλαδή να κάνουμε με την ιστορική αγορά και την συμβολή σε μια μελλοντική ανάπτυξη που θα ανταποκρίνεται πάνω απ' όλα στι ε, προσδοκίε των πολιτών και των επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δοθεί λοιπόν η έμφαση στην καινοτομία, τι θα πρέπει να κάνουμε στη σχέση με τα δικαιώματα του παραγωγού. Πώ μπορούμε να έχουμε και μια εσωτερική αγορά που λειτουργεί καλά, αλλά και διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μαλλών. Και από τι συζητήσει, οποίε διεξάγαμε μαζί και θα ήθελα να ευχαριστήσω προκειμένου όλου ε, και του συγκητέ, του συντάκτε των νομοδοτήσεων και όλου του συναδέλφου που διατύπωσαν τροπολογίε, μπορέσαμε να προσδιορίσουμε πέντε προτεραιότητε που θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Αμέσως. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω την υποστήριξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στην ιστορική αγορά, έτσι ώστε να έχουμε μια ισχυρότερη αλλά και πιο βιώσιμη ανάπτυξη, ένα νέο σύστημα ευρεσιτεχνίας και επίλυσης διαφορών που ήδη προχωρεί, ένα σύστημα, μια βελτιωμένη μάλλον προστασία των δικαιωμάτων του πνευματικού δημιουργού που έχουν τεράστια σημασία. Και αν θέλουμε την καινοτομία, θα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο χρηματοδότησή τη, όπω παραδείγμα τη μακροπρόθεσμε ε, επενδύσει και έναν τρόπο που θα επιτρέψει και στα κεφάλαια διακινδύνευση, κονδύλια, κεφάλαια να προχωρήσουν στι επενδύσει. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και επενδύσει ε, για τι ε, υποδομέ για τις τηλεπικοινωνίες με τις μεταφορές. Τρίτη προτεραιότητα είναι η ψηφιακή ε, ατζέντα στην ε, εσωτερική αγορά, δηλαδή ηλεκτρονικό εμπόριο, που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή αλλά και των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο με την καταπολέμηση και της πειρατείας και της απομίμησης προϊόντων και με τη διευκόλυνση ταυτόχρονα των, της μεταφοράς πέρα των σύνορων των προϊόντων. Το τέταρτο στοιχείο, σημείο αυτών των προτεραιοτήτων είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, με την ε, οικονομική του ανάπτυξη και τη δημιουργία των θέσεων εργασία που μπορούν να προσφέρουν χάρη σε μια ιστορική αγορά με φορολογικά μέτρα ε, ενσωματωμένα, ολοκληρωμένα ω προ το φόρο των επιχειρήσεων, με μείωση του, του γραφειοκρατικού φόρτου που θα επιτρέπει την αναπτύξη των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πέρα των συνάρων. Και πέμπτον, θα πρέπει να έχουμε εξορθολογισμό τη λειτουργία ε, των διαδικασιών αυτών για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν για να μπορούν να υποστηρίζουν ε, μια καλή, μια βιώσιμη, μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής τώρα ο κύριο Μπαρνιέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. κύριε και κύριοι βουλευτέ, βρισκόμαστε σε μια στιγμή κομβική σε αυτέ τι προσπάθειε που από κοινού ξεκινήσαμε υπό το φω της διαυγού και πλήρους εξέντασης τη εσωτερική αγορά από τον κύριο Μόντι με και υπό το φω τη της Grace που εγκρίνεται με μεγάλη προψηφία. Βρισκόμαστε επίση σε μια στιγμή που αν ακούσουμε καλά τους πολίτες της χώρα μας, διαπιστώνουμε ότι είναι καιρό να ξαναδούμε τη γραμμή του ορίζοντα για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη. Τι λόγια φεύγουν από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο στον κόσμο. Αναγκαίες αλλά δύσκολες, δεσμευτικές λέξεις πάντα. Ρύθμιση, δουλειά, διακυβέρνηση, εποπτεία, περιορισμός των ελλημάτων του χρέους, αναγκαία λόγια, δύσκολο τόσο και δεσμευτικά. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα και άλλες λέξεις, κυρίως άλλες δράσεις για να ξαναδώσουμε εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Τους λόγους δηλαδή για τους οποίους δουλεύουμε όλοι μαζί και όχι ο καθένας μόνος του για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Αυτό είναι τα θεμέλια των αιτιών της δουλειά μας. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την, τους εισηγητές σας, κυρία Καρνιέτη, κύριε Κοριέντε Κάμπος, τον κύριο Μπουσόη, να ευχαριστήσω τον κύριο Χάρμπο, αναφέρθηκε ήδη, με εξαιρετική αποτελεσματικότητα και κατανόηση επέτρεψε να προχωρήσουμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, σε όλες τις επιτροπές, να ευχαριστήσω επίσης και τους συντονιστές των διαφόρων πολιτικών ομάδων, διότι είχε πολλή δουλειά που έπρεπε να συντονιστεί μεταξύ σας. Ήταν πολλά τα ζητήματα που μας απασχόλησαν. Πιστεύω ότι αν προχωρήσουν τα πράγματα σωστά θα δώσετε και ένα πολύ καλό μήνυμα και στους άλλους ε, θεσμούς αλλά και στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Υπό το φως των εκθέσεων Μόντι και Γκρέσ, ο κύριος Μπαρόζο μου ζήτησε να συνεργαστώ με 12, συνεργά, με 12 επιτρόπους για την μεταρρύθμιση τη εσωτερική αγορά, τι διαθροτικέ μεταρρυθμίσει που θα επιτρέπουν να βρούμε 2, 3, 5 σημεία ανάπτυξης μέσα σε αυτήν. Και σα υπενθυμίζω κύριε και κύριοι βουλευτέ, ότι σε αυτή τη μεγάλη αγορά που είναι η πρώτη φάση του ευρωπαϊκού πολιτικού εγχειρήματο άλλωστε, 60% των εξαγωγών μα πηγαίνουν προ τι υπόλοιπε 26 χώρε τη Ένωση. Κάθε χώρα από τη Γερμανία μέχρι τη μικρότερη χώρα, 60% των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων της, της τα εξάγει δίπλα. Άρα η καλύτερη, εργασία, η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Εξού και η διαμόρφωση του Single Market Act και οι 50 προτάσεις που περιλαμβάνουν σε αυτό το μικρό μπλε βιβλίο που έστειλα σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις χώρες, σε όλους τους εθνικούς βουλευτές, τα συνδικάτα, τις επαγγελματικές οργανώσεις. Επίσης, ασχοληθήκαμε παρκώς με την συζήτηση για να επιλέξουμε μεταξύ των προτάσεων αυτών εκείνες που θα ήταν πιο αποτελεσματικέ για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων. Και την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη συγκεκριμένα, θα συζητηθεί στο Κολέγιο των Επιτρόπων το Single Market Act και μετά τις δικές σας συζητήσεις και αποφάσεις θα λάβει τα αναγκαία μέτρα. Για να κερδίσουμε κυρίε και κύριοι τον αγώνα της ανταγωνιστικότητας χρειαζόμαστε κάθε έδαφος, κάθε επιχείρηση, κάθε πολίτη, κάθε έδαφος. Γιατί στο ξεκίνημα της ενιαίας αγοράς και της ενιαίας πράξης η βούληση του Ζακ Τελόρ, πρόεδρου της Επιτροπής τότε, ήταν ακριβώς να συνοδευτεί η ενιαία αγορά με μια πολιτική συνοχής. Ούτως ώστε οι περιφέρειες που είχαν η στέρηση στην ανάπτυξη να μπορούν και αυτές να προχωρήσουν στη μάχη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Κάθε περιφέρεια της Ένωσης, ακόμα και οι ακραίες οι περιφερειακές περιοχές. Κάθε επιχείρηση έλεγα είναι αναγκαία. Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε παραδείγματο χάρη τα διπλώματα ευρεσιτεχνία που θέλουμε να προχωρήσουμε. Όταν θέλουμε να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να έχουν καλύτερη χρηματοδότηση, μικρότερο διοικητικό άχθο, να κάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο, να υπάρξει εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, να μπορούν να μετέχουν στις δημόσιες προμήθειες, το οποίο θα επανέλθω σε λίγο. Κάθε, κάθε έδαφος, κάθε επιχείρηση, κάθε πολίτης στην καθημερινότητά μας είμαστε όλοι καταναλωτές, χρήστες υπηρεσιών, αποταμιευτές, μέτοχοι, εργαζόμενοι, βιοτέχνες ο στόχος είναι να μπορούμε να διευκολύνουμε την κινητικότητα πέρα από τα σύνορα. Τα επαγγελματικά προσόντα, τα κοινωνικά δικαιώματα αυτών των ανθρώπων πρέπει να προστατεύονται και να αναγνωρίζονται, να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες ασφάλειας, να υπάρχει ασφάλεια όταν αγοράζετε προϊόντα υπηρεσίες από το ίντερνετ να μην υπάρχει διπλή φορολόγηση. Να κάποια παραδείγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να λειτουργήσει καλύτερη η εσωτερική αγορά. Ποιε είναι οι, συνέ... οι επόμενες φάσεις των συζητήσεων. Το εγχείρημα αυτό που έχουμε ξεκινήσει υπό μορφή συνομοθετικής διαδικασίας θα πρέπει να μας οδηγήσει στην επιλογή προτεραιοτήτων και όπως είπα ήδη την επόμενη εβδομάδα μαζί με τους συναδέλφους που είναι, με τους οποίους συνεργάστηκα πολύ στενά και τους ευχαριστώ θα προτείνω στο κολέγιο των επιτρόπων να επιλέξουμε 12 μοχλούς που θα επιτρέψουν να λειτουργήσει καλύτερα η εσωτερική αγορά. Κάθε μοχλός, κινητικότητα, χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων, πνευματική ιδιοκτησία, φορολογία, δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική συνοχή, Κάθε μοχλός έλεγα θα περιλαμβάνει μία κομβική δράση που θα είναι νέα, αποτελεσματική ελπίζουμε και για τις επιχειρήσεις και για τον πολίτη και παραδοτέα σε δύο έτη. Τι θα πει παραδοτέα. Την προτείνει η Επιτροπή και εσείς με το Συμβούλιο μπορείτε να λάβετε θέση και να εγκρίνει το κείμενο φέτος και του χρόνου. Μέχρι το 2012, μην ξεχνάτε, είναι τα 20 χρόνια της ε, ενιαίας αγοράς. Δεν έχουμε το δικαίωμα κυρίες και κύριοι, αν ακούμε καλά τι λένε οι λαοί της Ευρώπης, να αφήσουμε αυτή την επέτειο να γίνει μια νοσταλγική, μελαγχολική επέτειος. Πρέπει η επέτειος αυτή να είναι δυναμική για την ανάπτυξη. Έτσι θέλουμε να τη γιορτάσουμε μέσω του Single Market Act. 12 μοχλοί, 12 προτάσεις συγκεκριμένες, όχι όμως αποκλείουσες η μία την άλλη. Για κάθε μοχλό βρήκαμε και άλλες ιδέες, άλλες προτάσεις, άλλες δράσεις που θα προχωρήσει παράλληλα η Επιτροπή. Αλλά έχουμε 12 δράσεις κομβικές που θα είναι το σύμβολο όλου αυτού του εγχειρήματο. και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών, εσείς, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή από την πλευρά μας, η Ουγγρική Προεδρία που ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδίω την κυρία Υπουργό για την ε, αποφασιστικότητα με την οποία δεσμεύτηκε στο ζήτημα αυτό, επίσημα πριν τον Ιούνιο-Ιούλιο να αναλάβουν δέσμευση για να ε, προχωρήσει, να αποδώσει αυτό το Single Market Act. Αυτά ήθελα να σας πω. Μέσω μιας, μου ζητήσατε να αναφερθώ σε μία από τις διαστάσεις μέσω δήλωση επιτροπής. Να το κάνω τώρα για να αφήσω μετά το χρόνο στη συζήτηση. Περιλαμβάνεται στο Single Market Act και ενδιαφέρει το 17% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι δημόσιες συμβάσεις και οι δημόσιες προμήθειες. Να πω και εγώ δύο λόγια για τα τέσσερα εργοτάξια που έχουμε ξεκινήσει μαζί σας στον τομέα αυτό. Πρώτο μεγάλο έργο, η γενική αναθεώρηση της οδηγίας του 2004 για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των δημοσίων πόρων, για να επιτρέψουμε σε όσο περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται να μετάσχουν στις δημόσιες προμήθειες και να επιτρέψουμε την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με μικρότερη γραφειοκρατία. Συγκεκριμένα θέλω να απλοποιηθεί η διαδικασία, να γίνει πιο ευέλικτη, να δούμε πώς μπορούμε να λάβουμε καλύτερα υπόψη τις ειδικέ ανάγκες των μικρών τοπικών αυτοδιοικήσεων φερειπίν μέσω απλοποιημένων διαδικασιών. Δεύτερον, να διευκολύνουμε την ε, πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες μέσω κυρίως της διασυνοριακής συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τρίτον, να ενθαρρύνουμε, όπως ε, το ζήτησε ο κ. Χάρμπορ, με τον αλφα-β τρόπο πιο υπεύθυνε οικολογικές πράσινες αγορές που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την κοινωνική ένταξη. Οι στόχοι της μεταρρύθμισης θα γίνουν τώρα απλοί και πιο ισορροπημένοι κανόνες. Ξεκινήσαμε χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει μια μεγάλη διαβούλευση και οικονομική αξιολόγηση επιτόπου. Έχουμε μια πράσινη βίβλο και θέλουμε αυτή τη στιγμή να βρούμε τις πιο λειτουργικές δραστηριότητες. Δεν θα γίνουν παντού νομοθετικές παρεμβάσεις. Θα παρέμβουμε και με κλαδικές ε, παρεμβάσεις, καλύτερης χρήσης των δημοσίων ε, συμβάσεων, ενθάρρυνση στρατηγικών που περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, ενημέρωση φερρυπίν του εγχειριδίου για, μια, για οικολογική ε, για οικολογικές αγορές, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου οικολογικής αποτελεσματικότητας, επίδοσης, ενθάρρυνση του έργου αγορά καινοτόμων αγορών πριν τη θέση του εμπόριο σε συνεργασία με τον ε, κύριο και την κυρία Κουίν. Αυτό είναι το πρώτο εγχείρημα. Το δεύτερο είναι οι άδειε. Περιμένουμε ούτως ή άλλως αυτό το μακρόπνο έργο αναθεώρησης ε, της, ε, των δημοσίων συμβάσεων, αλλά θέλω να μιλήσω για τις άδειε. Οι άδειε, κυρίε και κύριοι, παίζουν ένα όλο και σημαντικότερο ρόλο στην παροχή υπηρεσιών δημοσίου χαρακτήρα. Το 60% των ΣΒΙΤ, των ε, συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη, γίνονται μέσω παραχωρήσεων. Παραχωρήσεων έργου κυρίω. Αυτή τη στιγμή ωστόσο δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία για τι παραχωρήσει. Παρότι εφαρμόζονται και σε αυτέ οι γενικέ αρχέ τη συνθήκη, υπάρχει στον τομέα αυτό μία ε, μικρή ασφάλεια δικαίου που επιβαρύνει τι συμβάσει αυτέ. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξαν 24 αποφάσεις του δικαστηρίου σχετικά τα τελευταία χρόνια. Θα προτείνω λοιπόν τη δημιουργία ενός περιορισμένου ελαφρού πλαισίου με κάποιους βασικούς κανόνες που δεν θα αμφισβητεί το εθνικό ε, κανονιστικό πλαίσιο όταν αυτό λειτουργεί καλά, δεν θα επιβάλλει υπερβολικό διοικητικό βάρος στην, ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίω λόγω των κατοφλίων που θα προτείνω. Ξέρω ότι υπάρχουν επιφυλάξει, υπάρχουν συζητήσει στι ομάδε για το θέμα αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένο, ακούγοντα όλου σα, ότι αν θέσουμε σωστά του στόχου, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τι παρανοήσει οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι ελεύθερες να οργανώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, να τις αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να τηρήσουν κάποια μίνιμουμ διαφάνειες και κανόνες που θα εξασφαλίζουν μη διάκριση. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη κατά άποψή μου για την καλύτερη χρήση των δημοσίων πόρων και τη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης χωρίς δυνατότητες προσφυγής αλλά και να μειωθεί η διαφθορά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επιχειρήσεις θέλουμε να ενσωματώ, να βελτιώσουμε την ε, εσωτερική αγορά. Άρα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την έννοια των παραχωρήσεων ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα δεν έχουν τα μέσα που διαθέτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις για να εξασφαλίσουν μεγάλες ε, συμβάσεις στις αγορές εάν δεν έχουν κάποια μορφή ε, παρουσίας και άρα χρειάζεται να διευκολύνουμε την ε, πρόσβαση των ε, μικρών επιχειρήσεων στις αγορές. Έχουμε επίσης και ζήτημα με την βελτίωση των ρυθμιστικών μέτρων, δηλαδή μία λύση που πιστεύουμε θα λύσει θα μα βοηθήσει να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα από ότι άλλε νομοθετικέ παρεμβάσει. Επίση, ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό τη ιστορική αγορά τη άμυνα. Για να προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα, θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για θέση εφαρμογή τη οδηγία του 2009, τη οποία η προθεσμία για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία ε, εκπνέει σε μερικέ εβδομάδε. Έχουμε να κάνουμε με ε, αντισταθμίσεις οι οποίες μερικές φορές είναι και αντίθετες ευθέως στο ευρωπαϊκό δίκαιο και θα ήθελα επίσης να συνεργαστώ με τον κύριο Ταγιάννη για το θέμα αυτό σε μια διάσκεψη που θα γίνει στα κτίρια του Κοινοβουλίου 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα επίση να υπενθυμίσω ένα θέμα το οποίο παραγνωρίστηκε για αρκετό καιρό, τη διεθνή δηλαδή διάσταση των δημοσίων ε, προμηθειών των αγορών. Είναι σαφής ο στόχος, περισσότερη πρόσβαση δηλαδή στον, στις αγορές αυτές για τις επιχειρήσεις μας και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε ακόμη περισσότερη βοήθεια μέσα σε ένα πνεύμα και αμοιβαιότητα βέβαια, αλλά και αμοιβαίων ε, συμφερόντων στο πνεύμα του «more trade will benefit all», περισσότερο εμπόριο προ το καλό των πάντων. Ε, με βάση αυτό όμω το αξίωμα του ανοιχτού εμπορίου και του, των πλέον εκτιμάτων προκύπτουν ε, εξ αυτού, αντιμετωπίσουμε το εξή πρόβλημα και θα το υπενθυμίζω ότι στην πραγματικότητα δηλαδή οι κύριοι εταίροι μας, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία στο πλαίσιο του GPA, η Κίνα σε διμερές επίπεδο, δεν θέλουν στην πραγματικότητα να δεσμευθούν και να ανοίξουν περισσότερο τις αγορές τους. Και εμεί από πλευρά μα δεν έχουμε πραγματικό μοχλό για να πιέσουμε στι διαπραγματεύσει στο βαθμό που οι δικέ μα οι αγορέ ήδη θεωρούνται σχεδόν ε, ω εκφύσεω ανοιχτέ αγορέ. Με βάση λοιπόν ε, τις ε, αρχές της Συμφωνίας Γενικών Γενικευμένων Προτιμήσεων ή του Παγκόσμιου Μηχανισμού Εμπορίου υπάρχουν κανόνες κυρίες και κύριοι που δεν έχουν εφαρμοστεί από αυτούς τους εταίρους και <clears throat> αυτό βέβαια σημαίνει Στρεβλώσει και για την εσωτερική αγορά. Οι δικές μας επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις ευρωπαϊκές αντιμετωπίζουν αυτή την άνηση κατάσταση πολλές φορές προβλήματα όπως αυτά των αυτοκινητοδρόμων της Πολωνίας Φερρυπίν με τη δυνατότητα για ορισμένους εταίρους να έχουν πρόσβαση στις δικές μας αγορές πολύ πιο προωθημένες από ό,τι έχει διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αφετέρου δε οι δικές μας επιχειρήσεις όταν θέλουν να βγουν στο εξωτερικό και να συμμετάσχουν στις αγορές ορισμένων εκ των μεγάλων μας εταίρων αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Γι' αυτό προτείνεται εφέτος ένα νομοθετικό μέτρο με τον κύριο Ντεκιούχτ, κυρίως τον συνάδελφο, που θα μετατρέψει σε ευρωπαϊκό δίκαιο τις δικές μας διεθνείς υποχρεώσεις σε θέματα ε, δημοσίων αγορών και θα μας δώσει και το μέσο μόχλευσης για τις διαπραγματεύσεις που χρειαζόμαστε. Εμείς είμαστε ναι υπέρ του ε, ανοιχτού εμπορίου, ε, του ελεύθερου εμπορίου, αλλά δεν είμαστε και ε, αφελείς. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να διαπραγματευτούμε μαζί με τις χώρες εταίρους συμφωνία για την οποία θα με την οποία θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη ε, ασφάλεια και για τις επιχειρήσεις μας. Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε βέβαια την Ευρώπη σε ένα φρούριο, αλλά θέλουμε οι επιχειρήσεις μας να έχουν και ρεαλιστικό και ισότιμο πεδίο δράσης σε ένα εμπόριο, όπως είπα, ελεύθερο, αλλά όχι σε όρους αφέλειας. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε, ιδιαίτερω για την επαναπροώθηση τη εσωτερική αγορά, για το σημαντικό αυτό τομέα που θα αποτελέσει άλλωστε κομμάτι αυτών των 12 μοχλών, στου οποίου αναφέρθηκα νωρίτερα, των ε, δημοσίων αγορών, του εξυγχρονισμού. Τα θέματα δηλαδή που θα μα περιμένουν και τι επόμενε εβδομάδε συζητήσει μα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. θα ακολουθήσει η Υπουργός κυρία Γιώρη εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Όπως ελέγχθη ήδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται μια κινητήρια δύναμη για την οικονομία της. Αυτό είναι το όραμά μας. Σας υπενθυμίζω ότι ήδη στην αρχή της Ουγγρικής Προεδρίας είχαμε πει καθαρά ότι το θέμα το βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν αρκεί δηλαδή να εγκύψουμε μονάχα σε μια προσπάθεια λύσης για την κρίση. Χρειάζεται να δώσουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να εξοπλίσουμε τις χώρες μέλη, υπάρχουν και διάφορες νομικές διατάξεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε, ώστε σε σχέση με το πακέτο αυτό να γίνει και η διαχείριση της κρίσης, αλλά Παραμένοντα ανταγωνιστικοί. Αυτό μπορεί να γίνει μονάχα εφόσον δημιουργηθούν νέε θέσει απασχόληση. Αυτό είναι και το σημαντικότερο από όλα. Αλλά χρειαζόμαστε και τι αντίστοιχε πηγέ. Πώ θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είμαι πεπισμένη ότι η ενιαία αγορά μα προσφέρει μια μεγαλειώδη ευκαιρία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και εδώ μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα σε συνδυασμό και με τη στρατηγική μας της Ευρώπης του 2020. Εκφράζω λοιπόν την ικανοποίησή μου για την δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της ενιαίας αγοράς. Είμαστε σύμφωνοι με τις προτεραιότητες που εκφράζονται και στις εκθέσεις σας και με τις οποίες συμφωνούν και οι άλλες δύο πλευρές. Ήδη υπήρξε η έκθεση του Λουί Γκρέσ που αποτέλεσε την βάση για επικοδομητική ανταλλαγή σκέψεων και εμείς τα υποστηρίζουμε αυτά. Έχουμε τώρα τις τρεις εκθέσεις. Έχουμε μια στοχευμένη συζήτηση που πρέπει να διεξαγάγουμε και ελπίζουμε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Ο Επίτροπος κ. Μπαρνίε είπε ήδη ότι θέλουμε να μπορέσουμε να εορτάσουμε με ενθουσιώδη τρόπο την επέτειο της ε, ενιαίας αγοράς. Ήδη το Συμβούλιο έχει εγκύψει τα κριτήρια που είναι απαραίτητο να θεσπιστούν για τους κατά προτεραιότητα τομείς και που πρέπει να υιοθετηθούν από τα θεσμικά όργανα και από τις χώρες μέλη. Και είδαμε ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός δέσμευσης από όλες τις πλευρές. Η Ουγγρική Προεδρία έχει άλλωστε τονίσει κατά επανάληψη ότι είναι σημαντικό αυτό. Στις 30 Μαΐου το Συμβούλιο θα ε, θα εγκρίνει τα σχετικά πορίσματα και θα κάνει τις σχετικές ε, θα δώσει μάλλον τις σχετικές κατευθύνσεις. Επιτρέψτε μου σύντομα να έρθω στο πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζουμε. Βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσης και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και ε, τα θεσμικά όργανα δεν βλέπουν πλέον να έχει ιδιαίτερη προστεθέμενη αξία η ε, αγορά. Το είπε και ο καθηγητής Μόντι. Αλλά είπε ότι πρέπει ειδικά σε αυτή, τέτοια, μέσα σε τέτοια περίοδο να υλοποιηθεί η ενιαία αγορά, διότι αυτή μπορεί να προσφέρει κίνητρα. Είμαι πεπισμένη ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε ένα πνεύμα απεσιοδοξίας. Πρέπει να προχωρήσουμε την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Είναι σημαντικό να βάλουμε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας τον πολίτη. Το είπαν ήδη οι βουλευτές σας. Αυτό άλλωστε διαλαμβάνει και η έκθεση Μόντι. Για την ώρα η ενιαία αγορά βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Εμείς πρέπει να εξαλείψουμε κάθε κόλλημα για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις βέβαια. Οι απαντήσει θα εξαρτηθούν πόσο, από το πόσο σημαντική είναι η δέσμευση από όλε τις πλευρέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα θα εγκρίνει την θέση του. Μέσα Απριλίου θα υποβάλουμε εμείς ανακοίνωση. Οι εκθέσεις σας αποτελούν και για μας κατευθυντήρια γραμμή. Αναμένουμε να δημιουργηθούν συνεργασίες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα που να επιτρέψουν την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς και να μπορέσουν να γίνουν και σχετικές επανεξετάσεις. Τώρα, θα έρθω με λίγα λόγια στις τρεις εκθέσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν θα επισέλθω βέβαια σε όλες τις λεπτομέρειες. Ως Προεδρία πάντως εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι ξανατίθεται επιτάπητος το θέμα της ενιαίας αγοράς. Εμείς θεωρούμε ότι η δέσμη αυτή μέτρων της ενιαίας αγοράς είναι καλή. Πρέπει να βρούμε τους σωστούς προσανατολισμούς και αυτό είναι βεβαίως καθήκον πρωτίστως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βεβαίως θα καθορίσει την ημερήσια διάταξή του. Τον Μάρτιο όμως ήδη συζητήσαμε σχετικά στο Συμβούλιο και ευχαριστούμε πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που μας έδωσε και αναμένουμε η υποστήριξη αυτή να συνεχιστεί και για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ένα συνολικό ενιαίο πλαίσιο ρυθμίσεων και αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία του γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μαζί του. Η ενιαία επίσης ψηφιακή αγορά είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση γιατί θα οδηγήσει σε ενίσχυση των επιχειρήσεων και εδώ πρέπει να προχωρήσουμε για παράδειγμα, στην καινοτομία, για παράδειγμα, στην κινητικότητα των πολιτών. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Έχουν τεθεί σημαντικά ερωτήματα. Χρειαζόμαστε ασφαλώς ενισχυμένη συνεργασία και αυτό είναι πρώτο στο καθήκον για όλους μας. Οι τρεις εκθέσεις που έχουν υποβληθεί ξεπηδούν κατά κάποιο τρόπο από την έκθεση Γκρέσ και τονίζουν ότι είναι απαραίτητο να μπει στο επίκεντρο των προσπαθειών ο πολίτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα. Υπάρχουν διάφορα, διάφοροι τομείς που μπορούν να ενισχυθούν, όπως για παράδειγμα το σύστημα Solvit, θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των πολιτών. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες προτεραιότητες τις οποίες έχει επιλέξει η Ουγγρική Προεδρία. Έχουμε προβλέψει και διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο. Βεβαίως μας έχουν ασκήσει κριτική και οι χώρες μέλη. Κριτική δηλαδή έχουν ασκήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διότι θεωρούν ότι δεν είναι, ε, δεν είναι εξασφαλισμένη η μακροοικονομική βεβαιότητα. Αυτό είναι σημαντικός στόχος που πρέπει να επιδιώξουμε και εντάσσεται και η στρατηγική μας της Ευρώπης 2020. Στην αρχή της ομιλίας μου τόνισα ότι η ενιαία αγορά προσφέρει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, το οποίο δεν επιτρέπεται να χάσουμε. Είναι σημαντικό για την ισορροπία ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διάφορα καθήκοντα τα οποία οφείλουμε να αναλάβουμε. Με τρόπο διαφανή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως θα συμμετάσχει στην προσπάθεια και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει και ελπίζει σε μια πλήρη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. έτσι Έχουμε τώρα τις πέντε παρεμβάσεις των τριών εισηγητών, του κύριου Επιτρόπου, της ε, εκπροσώπου του Συμβουλίου που δίνουν το ανακτήριο λάκτισμα για την συζήτηση. Για την εσωτερική αγορά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ανανέωση της εσωτερικής αγοράς είναι μια ιδέα που ξεκινά από την Επιτροπή των Οικονομικών την Επιτροπή Εσωτερική Αγορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Μάλκον Χάρμπορ και την Επιτροπή του που έδωσε την όθηση σε αυτήν την ε, ιδέα μέσα από την ε, έκθεση βέβαια του κύριου Μόντι. Ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Μπαρνιέ, τον Επίτροπο, για την ε, Εξαίρετη παρουσίαση και τόσο διεξοδική. και την παραπομπή στις δημόσιες αγορές που είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει στη πράξη. Η Ουγγρική Προεδρία ασφαλώς θα ασχοληθεί και εκείνη από πλευρά της έχει τεράστια σημασία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε πολύ σημαντικές εκθέσεις. Μια πολύ, σημαντική συζήτηση. Και αυτό το αποδεικνύει και ο αριθμός των επιτροπών του Κοινοβουλίου που έχουν ζητήσει ε, παρεμβάσεις στη συζήτηση αυτή. Έχουμε οκτώ συνολικά. Πολύ σπάνιο φαινόμενο να ζητούν τόσο πολλές ε, ε, επιτροπές στο λόγο. Θα παρακαλέσω λοιπόν τώρα την κυρία Αντρές Μπαρέα πρώτα, η οποία ομιλεί εκ μέρους της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οκτώ επιτροπέ ασχολήθηκαν, μία από αυτέ είναι η ΙΝΤΑ και ευχαριστώ τα μέλη τη επιτροπή μου για τι συνεισφορέ στην έκθεση. Η παγίωση τη εσωτερική αγορά είναι ένα ε, στόχο βασικό τη Στρατηγική 2020. Η ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο διεθνή πρωταγωνιστή ε, σε αυτόν τον τομέα και σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωση τι προκλήσει Σε προκλήσει για τι επιχειρήσει προκλήσεις στην διεθνή αγορά που περιλαμβάνει μεγάλες προσδοκίες και παρέχει πολλές ευκαιρίες αλλά και, ένα, μια διάσταση κοινωνικής ευθύνης, κοινωνικής ανάπτυξης με εγγυήσει για τους εργαζόμενους ε, και για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τις αναπτυσσόμενες χώρες ταυτόχρονα με δεσμεύσεις για τη μάχη κατά της φτώχεια, στόχους της χιλιετίας. Πρέπει να βοηθήσουμε τι επιχειρήσει να ενταχθούν στο μέλλον, στην γνώση του μέλλοντο, στον τομέα τη πνευματική ιδιοκτησία, στον αγώνα κατά των απομιμήσεων, να προσπίσουμε τι επιχειρήσει μα με βάση κριτήρια έρευνα και ανάπτυξη και κοινωνικά κριτήρια, καθώ και την εξωτερική διάσταση για του Ευρωπαίου πολίτε και του πολίτε εκτό Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Pan Diogo Feio, Komisja Gospodarcza i Κύριο κύριος Φέιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ καθώς και την Προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και βεβαίως ιδίως τους συναδέλφους της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής που συνεργάστηκαν για τις εκθέσεις. Όλα αυτά μου θυμίζουν πράγματι το πνεύμα της εκθέσεως του καθηγητού Μόντι όπου η ανταγωνιστικότητα μιας καινοτόμου αγοράς ε, τονίζεται με ιδιαίτερο τρόπο. Η στρατηγική Ευρώπης 2020 δεν πρέπει να μείνει ένα κενό κέλυφος. Δεν μπορεί να μείνει στα λόγια. Πρέπει να αποφέρει και πράξεις. υπέρ της ευρωπαϊκής οικονομίας. Χρειαζόμαστε μέτρα για να επιτρέψουμε την βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας με μέτρα τα οποία θα αποδώσουν και να επιτρέψουν μια πραγματική αύξηση της οικονομίας. Ο κύριος, Ο κύριος Μπαλτασάρε, ευχαριστώ πρόεδρε. Η σπουδαιότητα του Single Market Act βρίσκεται στο ότι θέλει να δώσει απαντήσεις στις απαιτήσει τη εσωτερική αγορά, διευκολύνοντα την πρόσβαση και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επιχειρήσεων, καταναλωτών και εργαζομένων. Έναντι του στόχου, του φιλόδοξου αυτού στόχου, θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικέ οι παρεμβάσει που πρότεινε ο κ. Μπαρνιέ και οι θέσει του Κοινοβουλίου. Κατά την άποψή μου, είναι επιτακτικέ κάποιε προτεραιότητε για να πετύχουμε του στόχου τη Ένωση. Ιδίω η βελτίωση τη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά ή με τη μείωση των διοικητικών υποχρεώσεων και με τη διευκόλυνση τη συμμετοχή του, στις διαδικασίες διαγωνισμών. Η κατάργηση κάθε εμποδίου στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η υποστήριξη και χρηματοδότηση τη κοινοτομία, ιδίω μέσω των εκπομπών ε, ομολογιών για έργα, ομολόγων συγγνώμη, για έργα της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών. Εν μόνο συνδέοντας την ανάπτυξη και τους, την υποστήριξη των επιχειρήσεων με τις στρατηγικές απασχόλησης της Ένωσης εν ώψη του 2020 θα μπορούσαμε να πετύχουμε τον στόχο της ενιαίας πράξης. Μια δημιουργία κοινωνική οικονομία της αγοράς που βασίζεται στην ανάπτυξη και την, και την βιωσιμότητα. Διακόπτεται ο μιλητής. Η κυρία Γιακονσάρη, Επιτροπή Απασχόλησης. Πρόεδρε, ο Ζακ όταν δήλωνε ότι η εσωτερική αγορά δεν θα γίνει αγαπητή, είχε άδικο. Το βλέπουμε αυτό από την συζήτηση. Είναι φιλόδοξη η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια προσέγγιση ε, η οποία περνάει μέσα από μεγαλόπνοα σχέδια. Κάτι ακόμη όμως που περιμένουμε είναι οι εκθέσεις να καλύψουν και θέματα που λείπουν ε, Φερρυπίν, το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική ρήτρα, την απόσπαση των εργαζομένων. Θέματα δηλαδή τα οποία δυστυχώ έχουν διατυπωθεί κατά πολύ γενικόλογο τρόπο. Και διρωτάται κανεί γιατί τα κοινωνικά δικαιώματα να θεωρούνται ω προβλήματα και δυσκολίες. Εγώ θα υπενθυμίσω στου αδέλφου ότι στι βόρειε χώρε, στις ε, χώρε ε, τη Σκανδιναβική, ε, έχουν συνδυαστεί τα κοινωνικά δικαιώματα με μεγάλη παραγωγικότητα και ε, καλές επιδόσεις στην οικοδομία. Δεν θα μπορούσατε κύριε Επίτροπε να δώσετε προσοχή και στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κρόιτσμαν από την Επιτροπή Απασχόληση επίση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα έλθω σε αυτό που είπε μόλι η συνάδελφο μου. Στην Επιτροπή μα, αντί για κοινωνική ρήτρα, προτείναμε να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των μέτρων της ενιαία αγορά στην απασχόληση. Αυτό βρίσκουμε ότι είναι πολύ σημαντικότερο από το να χρησιμοποιούμε κάποιες γενικές ρήσει. Να δούμε τα πράγματα που πρέπει να γίνουν στην ενιαία αγορά, τι επιφέρουν στον κοινωνικό τομέα. Και γι' αυτό χρειάζεται μια μελέτη επιπτώσεων που να λάβει υπόψη ακριβώ αυτά τα στοιχεία. Εγώ πάντως ευνηδιάστηκα όταν ο πρόεδρος της Economic Governance της κατεύθυνσης της οικονομίας δηλαδή, που δεν έχουμε εμείς καλές ε, εμπειρίες στη Γερμανία με τέτοιου είδους προσπάθειες. Θέλουν τώρα να τα βάλουν στην έννοια αγορά. Σωστό είναι να εναρμονιστούν οι οικονομίες μας, αλλά δεν θα βελτιώσουμε την ενιαία αγορά εάν προωθούμε την ιδέα της άνωθεν ρύθμισης της οικονομίας. Τα, επόμενο, το επόμενο έτος έχουμε βέβαια την 20η επέτειο της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό και χαίρομαι για τις δηλώσεις του Επιτρόφου Μπαρνίε που είπε ότι θα περιοριστεί σε ολίγα μόνο μέτρα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν επιβληθεί και τα οποία θα μπορέσουν να προσφέρουν νέα όθηση στην ενιαία αγορά η οποία ενιαία αγορά είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία για όλους μας μπορεί να προσφέρει περισσότερη απασχόληση και ιδίω των νέων. Αυτή είναι και η καλύτερη κοινωνική πολιτική που μπορούμε να ασκήσουμε. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε απασχόληση έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και την ίδια τους την προσωπικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να υποστηρίξουμε κάθε μέτρο το οποίο θα επιφέρει βελτίωση στην απασχόληση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ισορροπημένο πακέτο μέτρων το οποίο να προσφέρει πλεονεκτήματα και στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, ιδίω δε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε αυτές να μπορέσουν να υποφεληθούν περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα από την ενιαία αγορά. Θέλουμε επιτέλους το, η Ευρωπαϊκή Ευρεσιτεχνία, το δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας να είναι ε, προσιτό σε κόστος, ώστε να προστατεύει τις επιχειρήσεις. Θέλουμε και περισσότερα χρήματα να είναι διαθέσιμα για κεφάλαιο διακινδύνευσης, για risk capital και θέλουμε και ενιαία βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Από την άλλη μεριά θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ενιαία αγορά, να βελτιωθεί και η αναγνώριση προσόντων και επαγγελματικών ιδίως, γιατί με τον τρόπο αυτό προσφέρουμε και στους πολίτες και των δύο φίλων περισσότερη κινητικότητα μέσα στην ενιαία αγορά. Εκτός από αυτό χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή εποπτεία της αγοράς. Τονίζω, ευρωπαϊκή, διότι βλέπουμε συχνά οι χώρες μέλη να μην τα καταφέρνουν σωστά. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια... Σας ευχαριστώ, διακόπτει ο Πρόεδρος, τον κύριο Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεάντζελης από την Επιτροπή βιομηχανία. Έρευνα και ενέργεια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη προ την αγορά θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητε στι ανάγκε των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Πρέπει επίση να δοθεί μεγάλη προσοχή σε εγγυήσει κοινωνική διάσταση στην μελλοντική εσωτερική αγορά. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, των εργαζομένων και των χρηστών δημοσίων υπηρεσιών. Η ανάπτυξη, η και η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Μια οικονομική διάσταση προ όφελο των πολιτών. Το πακέτο κανόνων για τις επιχειρήσει περιλαμβάνει από την άποψη αυτή κάποιε καλές προτάσεις. Μεταξύ αυτών, το πρόγραμμα δράση για την αύξηση τη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κεφαλαία αγορά. Οι νέε γραμμέ χρηματοδότηση για καινοτόμε επιχειρήσει και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι η καρδιά τη οικονομία μα και ο κινητήρα ανάπτυξη εσωτερική αγορά. Δική μα ευθύνη, πρόεδρε, είναι να εξασφαλίσουμε του στόχου αυτού για να βγούμε από την κρίση και να ενθαρρύνουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξη βιώσιμο με, με απασχόληση ποιότητα. Ευχαριστώ η κυρία Σόφη Ακόνιε από την Περιφερειακή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα πράγμα θα να σας πω. Μια κουβέντα, μια κουβέντα που ίσως να ε, παρουσιάζει σημεία τομής με την τωρινή ε, συγκυρία, αλλά πάντως αποτελεί πηγή φιλοδοξίας φιλοδοξία για την Ευρώπη, για την εσωτερική αγορά, φιλοδοξία να δείξουμε στον πολίτη ότι έχει δικαίωμα και δικαιώματα και ως εργαζόμενος και ως καταναλωτής και ως ταξιδιώτης μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάνω απ' όλα ως ιδιώτης, ως άτομο πάνω απ' όλα. Και σε αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μισελ Μπαγνιέ για όλα τα μεγάλα και μεγαλόπνοα σχέδια που θέλει να ε, θέσει εφαρμογή ως συντάκτης νομοδότησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που ε, έχει στο και ό,τι στα θέματα τη περιφερειακή ανάπτυξη. Ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έμφαση που δίνεται στι περιφέρειες με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπω τι άκρω απομακρυσμένε περιφέρειε, την ιδέα μια ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία, του του καταστατικού μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης, της ε, έκδοσης ομολογιών για συγκεκριμένα σχέδια και του σχεδίου για την ανάπτυξη της, ε, για μια βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπιότρ Μπόρης έχει το λόγο τώρα. Πρόεδρε. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα εδώ πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για τους στόχους της ε, Ευρώπης για το 2020, καινοτομία δηλαδή, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία ε, σχετίζονται άμεσα με την εσωτερική αγορά και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Επίτροπο για την ε, παρουσία του εδώ για τα όσα είπε και για τη συνέχιση του έργου του κυρίου Μόντι. Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνία μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, ελπίζουμε, του χρόνου του 2012, δηλαδή, όπου θα χαιρετίζουμε και την 20 από την ε, θέσπιση της, ε, την ανακήρυξη μάλλον της εσωτερικής αγοράς, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο, ένα σύστημα για την ε, διαχείριση των δικαιωμάτων του παραγωγού, του πνευματικού δημιουργού και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απλούστευση των νομικών διατάξεων και των διαδικασιών, με την θέσπιση ενός καταστατικού, με ένα κοινό μητρό επιχειρήσεων, όπου θα μπορέσουν να βρουν ε, τη θέση τους σε 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος και παρακαλώ μην μιλάτε τόσο γρήγορα. Δεν είναι δυνατόν να μεταφραστείτε. Ο κύριος Λένε δεν είναι παρόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριος Μάντερς, από την Επιτροπή των Νομικών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Α, θα μου δώσετε λοιπόν το, τα λεπτά του κυρίου Λένε. Ευχαριστώ πάντως πρώτα πρώτα τον κύριο Επίτροπο καθώς και όλους και όλες που είναι παρόντες ή παρούσες εδώ. Ε, συζητήθηκαν εδώ ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα. Τα έχω βάλει και στο κείμενό μου εγώ. Ελπίζω να τα περιλάβει ο ο κύριος Επίτροπος στις σκέψεις του επενέθηκε πολύ η έκθεση του κύριου Μόντι που λέει όμως ότι χρειαζόμαστε και περισσότερα δικαιώματα για την ενιαία αγορά. Πρέπει να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση να αποφύγουμε αυτό το παζλ των 27 διαφορετικών ε, νομοθεσιών. Το πιο σημαντικό, πιο σημαντική παράληψη για μένα μέχρι τώρα είναι η έννοια του marketing. Έχουμε θαυμάσιους νομικούς, βελτιώνουμε την ενιαία αγορά ε, υπέρ του πολίτη, αλλά ο πολίτης δεν το αντιλαμβάνεται, διότι δεν υπάρχει η επικοινωνιακή αυτή γέφυρα με τον πολίτη. Και αυτό διότι χρησιμοποιούμε μοναχά νομική ορολογία και έχουμε μπροστά μας τον κίνδυνο να απομακρυνθούμε όλο και περισσότερο από τον μέσο πολίτη ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος ε, σε αυτό το θέμα στο μέλλον ώστε να προσελκύσουμε την προσοχή του πολίτη και να τον καταστήσουμε υποστηρικτή της ενιαίας αγοράς. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερους communication managers, ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό σωστά. Εξάλλου, ο Ευρωπαίος πολίτης εν τέλει δεν γνωρίζει την διάκριση, δεν ενδιαφέρεται για την διάκριση μεταξύ Ευρωβουλής, Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου ή ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας τα σκεφτούμε λίγο και αυτά. Ας φτιάξουμε έναν Ευρωπαίο πρέσβη, ο οποίος να μπορεί να δρά και να αντιδρά και να είναι ορατός. Διότι αλλιώς φοβούμε ότι μας αναμένει η μοίρα του Τιτανικού. Και εσείς, μιλήσατε. κάπως ε, γρήγορα, κύριε Μάντερς. Ο κύριος Βαντεκάμπ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο για τις ε, παρατηρήσεις του στην αρχή της συζητήσεως. Ξέρετε ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα την ε, τοποθέτηση και την γνωμοδότηση και της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών για, την, ε, για τις πολιτικές ελευθερίες. Νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ίδια την, ιδέα, την εσωτερική αγορά, πρέπει να υποστηρίξουμε της, ε, την εσωτερική αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών που έχει απόλυτα θεμελιώδη σημασία στην εσωτερική αγορά. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πολλοί και οι μετανάστε που διακινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να δώσουμε σημασία. Και πιστεύω ότι του επόμενου μήνε μαζί με τον κύριο Μπαρνιέ θα μπορέσουμε να δώσουμε νέα όθηση σε αυτά τα θέματα. Γιατί ο ανταγωνισμό δεν περιμένει. Πότε θα πάρουμε τι αποφάσει που μόνο του. Ευχαριστώ και καλημέρα. Ο κύριος Ματσόνη έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Η κυρία Ματσόνη, συγγνώμη. Πρόεδρε, επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κύριε Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι η δουλειά των εισηγητών είναι εξαιρετική. Είναι ιδιαίτερα δε θετικά τα λόγια της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Οι τρεις εκθέσεις διαφυλάσσουν το πνεύμα της ε, δυναμικής της ενιαίας αγοράς που περιλαμβάνεται στην έκθεση Μόντι και διαφυλάσσει την ενότητα του στόχου, την επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο μέσω 50 μέτρων που κατόπιν ε, επανεμφανίζονται συνθετικά στο Κοινοβούλιο με 14 προτεραιότητες. Στο εσωτερικό των μέτρων, μέσα από το μέτρο αυτό, 19 αφορούν την συγκέντρωση αγοράς στα συμφέροντα των πολιτών. Άρα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να πετύχουμε πλήρως την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς, μειώνοντας την απόκληση μεταξύ, την απόσταση μεταξύ πολιτών και αγοράς. Με μια δουλειά για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης των πολιτών στην εσωτερική αγορά μέσω της προώθησης διαδικασιών κοινωνικής και πολιτικής κυρίως και όχι οικονομικής ένταξης και μέσω μιας διαφορετικής θέσης της αντίληψης της εσωτερικής αγοράς για τους πολίτες της Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνονται στα μέτρα που βρίσκονται στις αυτές εκθέσεις. Ευχαριστώ. Εγώ, εγώ ευχαριστώ κύριε Ματσόνη. Αφού ακούσαμε την, τις ε, των επιτροπών θα προχωρήσουμε στου ατομικούς αγωγητέ. Ο κύριος Κάρας. Να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, μάθαμε ότι σήμερα το πρωί την Αυγή